Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. J'espère qu'il y aura de la place pour chacun. Λοιπόν, ελπίζω να χωρέσουμε. Και επαναλαμβάνω ότι οι εργασίες στις 2.30 όπως είχαμε πει ακριβώς. Οι τερμινείς σας ενημερώνουν ότι βρίσκονται στην 36η μέρα των κινητοποιήσεων κατά των συνθηκών εργασίας που μας επέβαλε η διοίκηση. Δεν θα παραχωρήσουμε υπέρβαση ωραρίου τη συγκεκριμένη συνεδρίαση και θα σταματήσουμε στις 5.30 ακριβώς. Ο Πρόεδρος, προχωρούμε στην παρουσία της μελέτης, της μελέτης με θέμα της ανάλυσης της εκτέλεσης των διαρθρωτικών ε, ε, ταμείων και των επενδυτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Φαμπιάν Γκάλ ε, που δέχτηκε να επιστρέψει και το απόγευμα γιατί ήταν το πρωί η παρουσίαση αυτή. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι θα αφιερώσουμε το πολύ 20 λεπτά στο συγκεκριμένο θέμα και μετά θα ανταλλάξουμε απόψεις για την άμυνα. Είναι το σημείο 13, εξού και η παρουσία της κυρίας Κλέρ Μούντι, γιατί την καλωσορίζω. Και χαίρομαι που τη βλέπω εδώ γιατί συμμετείχε και στην Επιτροπή Προπολογισμών στο παρελθόν και έχουμε άριστες αναμνήσεις. Έχουμε αναβάλει και μια ψηφοφορία, θυμίζω, για την μεταφορά πιστώσεων υπαριθμών 18 του 2018 χρειαζόμασταν περισσότερες ε, πληροφορίες, οπότε και θα ψηφίσουμε κατά τις 5 και 20. Έχουν μια ανακοίνωση να μας κάνουν οι διερμηνείς, οι οποίοι έχουν ε, έρθει να εργαστούν υπό επίταξη. Θα πρέπει να τελειώσουμε ακριβώς στις 5.30, αν θέλουμε να έχουμε και διερμηνία, λέει ο Πρόεδρος. Ah. Monsieur Depré, vous avez raison Μπράβο σα, κύριε Δεπρέ που το γιορτάζετε εκ των προτέρων, λέει ο πρόεδρο. Ο έρθει με σημαία του Βελγίου και κασκόλ τη Εθνική. Θα τα ξαναπούμε τα βράδυ, λέει ο Χαρείτε, χαρείτε τώρα που μπορείτε. Eh, Bien, ils ont fait leur déclaration j'entends rien. Euh, J'ai rien entendu. Bon. Λοιπόν, κύριε Γκάλ, θέλετε να συνεχίσετε από εκεί που είχατε σταματήσει σήμερα το πρωί, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να τελειώσω την παρουσίαση αυτή σήμερα το απόγευμα και θα επανέλθω στα αγγλικά. Είναι λίγο περίεργο γιατί αυτή τη στιγμή που μιλούμε για τους ε, λόγους καθυστερήσεων ε, στην πολιτική ε, συνοχής έχει καθυστερήσει και η παρουσίαση αυτής της μελέτης από κάποιο απρόβλεπτο γεγονό όπω συμβαίνει και ε, στην ε, περίπτωση του Ταμείου συνοχή. Ε, λέγαμε λοιπόν για τι προτάσει μέχρι το 2020. υπάρχουν ε, κάποια ωφέλη, Βεβαίω, αυτό θα πρέπει να το δούμε ε, κάπως σχετικά. Η ευελιξία είναι κάτι το ευπρόσδεκτο, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η πολιτική συνοχή ενέχει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και σχεδιασμό μπορεί να γίνουν αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα, τα λεγόμενα ΕΣΠΑ, τα οποία ε, μπορεί με τη σειρά τους να οδηγήσουν και αυτά σε καθυστερήσεις. Άρα, χρειάζεται ένας προγραμματισμός, ένας ε, σχεδιασμός και προγραμματισμός με απλούστευση. Πολλές φορές στο παρελθόν, πάρα πολλές φορές, έχουμε ακούσει εξαγγελίες για απλούστευση, για απλοποίηση των ε, διαδικασιών, αλλά στην εφαρμογή τους αυτά αποδείχτηκαν ακόμα πιο περίπλοκα. Άρα καλές οι προσπάθειες για την απλοποίηση, αλλά να γίνονται και πραγματικότητα. Επίσης, συνέργειες και συνοχή ε, χρειάζεται να προαχθούν. Αλλά στις προηγούμενες νομοθετικές προτάσεις εξαιρέθηκε το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου από τη δέσμη των μέτρων για τη συνοχή. Ε, πράγμα που δυσκολεύει τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Και τέλος, οι προσπάθειες που γίνονται να ε, περάσει νομοθεσία πριν τις ευρωεκλογέ. Ε, μπορεί να είναι κάτι θετικό, αλλά χρειάζεται να έχουμε και τον απαραίτητο χρόνο για να γίνεται ο σωστός κοινοβουλευτικός έλεγχος και οι συζητήσεις. Έρχομαι τώρα στα προβλήματα και τις προκλήσεις ε, της πρότασης. Οι διάφορες αρισιμότητες που έχουν αυξηθεί μπορεί να ε, επιβραδύνουν ακόμα και να σταματήσουν την εφαρμογή. Η μείωση της τεχνικής συνδρομής και βοήθειας ε, ενδεχομένω σημαίνει κόστος και βάρος διοικητικού και προσωπικού. Επίσης η μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης και οι προκαταβολές ε, εμπροστοβαρείς ε, πληρωμές μπορεί να προκαλέσουν κάποια προβλήματα ρευστότητα στα κράτη-μέλη. Επίσης, η μείωση του χρόνου διάρκεια νήση 3 έγινε νήση 2. Δηλαδή, ο χρόνος από τη στιγμή που δεσμεύονται τα κονδύλια μέχρι τη στιγμή που δαπανώνται έχει μειωθεί. Και αυτό μπορεί να ε, οδηγήσει σε προβλήματα όταν υπάρχουν αναπάντηχε καθυστερήσει η προσημείωση, αυτό το earmarking, ε, ότι ε, ορισμένα ποσοστά προσυπογράφονται για κάποιες θεματικές ενότητες και στόχους, μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες αυτά για κάποια κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη όπου έχουν αλλάξει ταξινόμηση οι περιφέρειες ε, ή έχουν πολλές περιφέρειες που είναι σε μεταβατική περίοδο. Για να κλείσω, μετά την καθυστερημένη έναρξη, η πολιτική συνοχή τώρα έχει μπει σε μια επιταχυμένη πορεία και υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη αλλά μεταξύ και των περιφερειών ίδιων κρατών μελών για διάφορους λόγους που συνδέονται με τη συνοχή και τα προγράμματα. Σε ένα ΕΣΠΑ μπορεί να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ε, για κάποιο λόγο που δεν προκαλεί καμία καθυστέρηση σε ένα άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάλογα με το κράτος μέλος. Ε, συνεχίζονται οι προσπάθειες σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ε, ξεπεραστούν τα προβλήματα και ε, πραγματικά οι προτάσεις για μετά το 2020 έχουν και θετικά και κάποια αρνητικά. Ε, συμπεράσματα και συστάσεις. Πρώτον, θα πρέπει να ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχουν οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία και πάντα να λαμβάνετε αυτό υπόψη. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει μια χάραξη προτεραιοτήτων και στόχων. Σε τι θέλουμε να επικεντρωθούμε, σε άκαμπτη δημοσιονομική πειθαρχία ή θέλουμε να αφήσουμε αρκετό χρόνο για την προετοιμασία, το στήσιμο, τη χάραξη στρατηγικής ε, να διδαχθούμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση είναι προσιλωμένη στην απλοποίηση και στην αναμόνιση. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η δημιουργία ικανοτήτων, αυτό το capacity building που πρέπει να συνεχιστεί και να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ε, την τεχνική βοήθεια σωστά και αυστηρά. Θα τελειώσω εδώ, σταματώ την παρουσίασή μου και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις θα είχατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Merci, Monsieur Gall. Merci. Ευχαριστώ κύριε Γκάλ για την παρουσίαση αυτής της μελέτης και τα συμπεράσματα όσο και τις συστάσεις σας. Απλούστευσε εναρμόνιση. Ευελιξία. Ανάγκη για τεχνική σύνδρομη και ελαστικότητα. Νομίζω οι δύο συνεισηγητές μπορούν να πάρουν το λόγο και να σας μεταφέρουν τις δικές τους απόψεις. Κυρία Τομά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις απόψεις σας. Θα ήθελα να αντιστέσω σε ένα άλλο ίσως λίγο πλαίσιο γιατί ήδη από την αρχή του ισχύοντος ε, πολιετούς δημοσιονομικού διαρωτώμεθα σύνεχως ε, για το χαμηλά ποσοστά κατανάλωσης των διαφορετικών ταμείων. Ακούγοντας την άποψή σας, φαίνεται ότι το ερώτημα αυτό δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένο, δικαιολογημένο. Εκφράζονται ανησυχίες όμως και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταλήγουμε πολλές φορές στο βιαστικό συμπέρασμα που λέει ότι τα ταμεία αυτά ίσως να μην είναι κατά κατάλληλα, δεν είναι σε σχέση με την πραγματικότητα και η προστιθέμενη αξία του αμφισβητείται. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χωρίς προκαταλήψεις αλλά με κάποιες αμφιβολίες γύρω από τους ισχυρισμούς αυτούς ζητήσαμε μία ανεξάρτητη μελέτη για την εφαρμογή των διαφορετικών ταμείων. Είπα χωρίς προκαταλήψεις για να κατανοήσουμε, για να διορθώσουμε. Γιατί τώρα για το επόμενο πολιετές θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι ε, προσαρμογές μπορούμε να κάνουμε Και θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με αυτά που μας λέτε, ακόμα και αν υπάρχει μια κάποια καθυστέρηση, τα ποσοστά απορρόφησης θα είναι αρκετά παρόμοια με αυτά τα οποία είχαμε ανάμεσα στο 2009 και το 2013 και γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο εγώ καταλήγω, στο οποίο καταλήγω, είναι ότι όποιος θέλει να σκοτώσει το σκύλο του λέει ότι είναι λυσασμένος. Συνεπώς λοιπόν η μη απορρόφηση και η μη χρήση των α, ταμείων αυτών δεν είναι κάτι το ακριβές. Τουλάχιστον στον βαθμό που θα μπορούσε να δικαιολογήσει αν δεν ήμασταν προσεκτικοί, στη μείωση των διαφορετικών ταμείων, κάτι το οποίο το Κοινοβούλιο δεν επιθυμεί. Η μελέτη σας στην ουσία ξεκαθαρίζει κάπως τα πράγματα και τώρα έχουμε πια συγκεκριμένες αιτίες αν θέλετε και συγκεκριμένες εξηγήσει για τα χαμηλά επίπεδα απορρόφησης στην αρχή της περίοδου στα θέματα τα σχετικά με την κρίση και να πω ότι δεν αναφερθήκατε στην κρίση. Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω ότι με δημοσιονομικά σοβαρά θέματα σε πολλές χώρες και με ε, πολλά θέματα επίσης σε επίπεδο δημοσιονομικών ελλημάτων υπάρχουν αρκετοί δισταγμοί να ε, δεχθούμε ε, δυνατότητες συγχρηματοδότησης λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν τουλάχιστον. Υπάρχει φυσικά και η διακανονιστική περιπλοκότητα. Η κυρία Γκρέσλε δεν είναι εδώ, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής Προϋπολογισμών να πω ότι το θέμα δεν είναι το Κοινοβούλιο να προσπαθήσει να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα ίσα ίσα κάθε δυνατότητα βελτίωσης της ε, διακυβέρνησης των, ε, των ε, θα έλεγα των συγκεκριμένων αυτών μέσων είναι κάτι που πρέπει να καλωσορίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σόλμπεστ. Νομίζω ότι μία φράση στην έκθεσή σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Στη σελίδα 9 μας λέτε ότι οι πληρωμές στα πλαίσια των προγραμμάτων 14 με 20 έρχονται ένα χρόνο αργότερα σε σχέση με το 2007-2013. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τις δύο αυτές δυνατότητες συγκρίνουμε ακριβώς την ίδια αντίστοιχα περίοδο, τρία με τέσσερα χρόνια, Το θέμα είναι να δούμε ποιο είναι το συμπέρασμα. Εμείς βρισκόμαστε στην ίδια περίοδο με τις ίδιες πληρωμές ένα χρόνο πιο ε, αργά. Έχουμε καθυστερήσει. Τι έχει συμβεί λοιπόν, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Εσείς μας δείξατε τις διαφορετικές συνθήκες που υπάρχουν εσωτερικές και εξωτερικές. Αυτές οι συνθήκες αναφέρονται και στην νομοθετική βάση και λυπάμαι που θα πω ότι αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ε, γιατί το Κοινοβούλιο συναποφάσισε. Θα ήθελα εδώ να ακούσω από τους ερευνητές ότι να μου πούνε ότι πραγματικά οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις είναι πολύ περίπλοκες. Και ακριβώς λόγω της περιπλοκότητας πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα για το 19 και 20, γιατί μένει ακόμα το 19 και 20. Τώρα για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Το σύστημα είναι πιο περίπλοκο λοιπόν από το 2007-2013. Το θέμα δεν είναι μία απλή γραμμική απλωστεύση, απλοποίηση. Πρέπει να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Τι γίνεται λοιπόν αν καθυστερήσουμε ένα, δύο ή τρία χρόνια όταν βλέπουμε όπως τώρα ότι καθυστερούμε. Αν δούμε ότι με το πολιετές δημοσιονομικό δεν είμαστε έτοιμοι πριν από τις εκλογές, οι αποφάσεις θα ληφθούν το 2020. Το σύστημα λοιπόν θα καθυστερήσει όχι ένα αλλά δύο μπορεί και τρία χρόνια. Τρία χρόνια καθυστέρηση. Γιατί γιατί το 21, 22 και 23 τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του προηγούμενου δημοσιονομικού. Γιατί με αυτό το ποσοστό απορρόφησης ε, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για παλαιού τύπου προγράμματα και ίσως να υπάρξει ένα κενό χρηματοδοτικό. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες πρακτικά της καθυστέρησης. Ποιες είναι οι συνέπειες της καθυστέρησης στη συνοχή. Αν δεν θα είμαστε έτοιμοι το 19 θα είμαστε έτοιμοι στο τέλος του 20. Τι συνέπειες θα υπάρξουν λοιπόν στην πολιτική συνοχή. Ίσως είναι ιδιαίτερα επίγον το θέμα αυτό γιατί για τις μεταβατικές περιόδους ε, ε, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τον ΙΣΕΝ 2 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μένει στον ΙΣΕΝ 2 και όχι στον ΙΣΕΝ 3. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή διότι μας δίνει ε, πληροφόρηση σε πραγματικά αριθμητικά στοιχεία. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά τον καθηγητή Μπάχλερ αλλά στο τέλος, ε, στα συμπεράσματά σας δεν είστε αρκετά αυστηροί και σκληροί. Είναι πιο πολιτικά και διπλωματικά συμπεράσματα. Ότι ναι, να δούμε. Όχι, τώρα θα πρέπει να βγουν σκληρά συμπεράσματα. Δηλαδή, ότι αν δεν είσαι έτοιμος ε, μέσα σε αυτό το διάστημα, να είσαι προετοιμασμένος και ότι θα κοπούν όλα. Τέτοιες προτάσεις θέλουμε, γιατί όταν μιλάμε εμείς για αυτά τα θέματα, μιλάμε σε άλλο επίπεδο από τους ειδικού που έχουν ε, τα στοιχεία. Λοιπόν, δεν έχουμε διαδικασία κάτσια για λόγους χρονικούς. Είδατε ότι αρχή το 2014-2015 ήταν πολύ αργή. Αναρωτηθήκατε πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί στις απαιτήσει πληρωμών δεδομένων των καθυστερήσεων των πληρωμών από την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, αν αρχίσουμε την 1η Ιουνίου 2021 ολοταχώς, η ιανουιου 2021 ολοταχως Επιτροπή θα έχει αρκετό ρευστό για να τα αντιμετωπίσει αυτά. Τρία λεπτά για να απαντήσετε στους δύο εισηγητές. Κύριε Γκά. Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω το συντομότερο. Και σε όσο γίνεται πιο σύντομο διάστημα. για την πολιτική συνοχής χρειάζεται μεγάλος χρόνος προετοιμασίας έτσι ώστε να αρχίσει να τη σε ισχύ. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Αλλά επίσης είδαμε ότι έγιναν και μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την προετοιμασία του. Αν δείτε αυτή τη διαφάνεια, στην αρχή αρχή στην ανάληψη υποχρεώσεων ήδη έχουμε καλύψει ε, τις καθυστερήσεις σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Και τι κάνουν οι διαχειριστικές αρχές, αν το μελετήσουμε, έχουν κάνει την προετοιμασία τους. Άρα αυτές οι καθυστερήσεις δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν προβλήματα τα επόμενα χρόνια, αλλά ε, μπορούν να υλοποιηθούν τα διάφορα έργα. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που εμπλέκονται για την περίοδο 2007-2013. Το νομοθετικό πακέτο δεν εγκρίθηκε όσο αργά υιοθετήθηκε το πακέτο του 2014-2020. Ωστόσο, για κάποιους λόγους θεωρήσουμε ότι ήταν καλό να το εξετάσουμε μετά από τέσσερα χρόνια. Και τώρα βρισκόμαστε ήδη τέσσερα χρόνια μέσα στη νέα περίοδο. Αυτό που συνέβη για την περίοδο 2014 με 2020 ίσως ένα παράδειγμα μιας διαδικασίας ήταν να έχουμε μια εύκολη άσκηση, μια... να περιγράψουμε τη δικασία στις ε, εκτελεστικές αρχές, αλλά στην πράξη είδαμε ότι αυτό οδήγησε σε ε, μακρές καθυστερήσεις, γιατί η περιγραφή έπρεπε να ε, εγκριθεί από την ελεγκτική αρχή, η οποία χρειαζόταν αποδείξεις. ότι τα, τα μέλη, οι εργαζόμενοι μπορούν να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά και ε, η ελληνική αρχή ζητούσε ε, ε ότι τα μέλη είχαν τις ικανότητες. Η διαχειριστική αρχή είπε λοιπόν ότι, ότι έπρεπε να έχουν επικαιρωμένα βιογραφικά για να μπορέσουν να το αποδείξουν αυτό ε, για παραπάνω από 20 χρόνια, ώστε να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να εφαρμόσουν ε, ε, τις πολιτικές. Έχω ξεπεράσει τα τρία λεπτά, οπότε ναι, θεωρώ ότι η καθυστέρηση στην έγκριση της νομοθεσία θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την περίοδο μετά το 2020. Συμφωνώ λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ ε, που δεχθήκατε να παρατείνετε ε, την ε, παρουσίαση σας και την παραμονή σας. Ευχαριστώ και τον συνάδελφό σας τον κύριο Φέρη και θα το αφήσουμε εδώ αυτό το θέμα για τα διαστατικά ταμεία και την πολιτική συνοχής. Προχωρούμε λοιπόν στην επόμενη ενότητα που αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμενας Με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, ο οποίους και καλωσορίζω, ιδιαίτερα την Αντιπρόεδρο Κλέρ Μούντι, η οποία επανέρχεται στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών, παλιό μέλος της θελήσαμε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για να καταλάβουμε καλύτερα τις σημερινέ και μελλοντικέ εξελίξεις μιας πολιτικής άκρος στρατηγικής που επιθυμούν και οι Ευρωπαίοι ε, πολίτες, που είναι η κοινή πολιτική Άμυνα και τι δυνατότητε χρηματοδότηση. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που αρχίζουν να λαμβάνουν σιγά σιγά σάρκα και οστά ή στο προσεχές μέλλον, η ΠΕΣΚΟ α πούμε διαρθρωμένη συνεργασία ή το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξη στην αμυντική βιομηχανία ε, όπου την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, έδωσε το η Ολομέλεια θα συζητηθούν και άλλα θέματα δημοσιονομικά με το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ή ε, η στρατιωτική κινητικότητα. Υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός του προεμπλογισμού της Ένωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα παραμείνει αδρανές απέναντι σε προτάσεις που δεν εντάσσονται στην συνήθι νομοθετική ε, διαδικασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μελλοντική κοινή ε, πολιτική άμυνας να είναι ε, στην υπηρεσία μιας πραγματικής στρατηγικής και πολιτικών επελογών. Και το Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων λοιπόν προαναγγέλει πάρα πολύ συναρπαστικές μελλοντικέ συζητήσεις. Για να διαρθρώσουμε τη συζήτησή μας, να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Πέντρο Σεράνο, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΕΙΕΔ, και μετά τον κύριο Σιλβάνο Πρέσα, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Χίλντε Χάρντεμαν, που είναι διευθύνουσα ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ε, Εξωτερικών Υπηρεσιών. Πριν του δώσω όμω το λόγο, να ακούσουμε την κυρία Κλέρ Μούντι από πλευράς υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ. Σα ευχαριστώ που οργανώσετε αυτή τη συνεδρίαση ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και πάλι μαζί σας. Είναι σαν να γυρίζω σπίτι μου να ευχαριστήσω και τους ομιλητές που είναι εδώ. Θα σας παρουσιάσουμε επισήμω σύντομα. Η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα είναι ένα τομέα που εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε δει νέα όθηση για πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, το νέο απειλητικό περιβάλλον στο οποίο ε, εργαζόμαστε και το οποίο απαιτεί περισσότερη και καλύτερη συνεργασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ως προς τη διευκόλυνση της εργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, πολύ σχετικό και με την Επιτροπή Προπολογισμών είναι ότι χρειάζονται καλύτεροι μηχανισμοί ε, δαπανών. Αυτό θα συζητήσουμε. Γνωρίζουμε ότι οι δαπάνες αντιστοιχούν στο 1,3% του ΑΕΠ ή σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ για 28 κράτη-μέλη. Το 2016 αυτό το νούμερο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο γιατί 22 κράτη-μέλη είναι παράλληλα μέλη του ΝΑΤΟ και ε, υποσχέθηκαν να αυξάσουν κατά 2% ε, τα έξοδα τους μέχρι το 2024. Βλέπουμε όμως και σε εθνικό επίπεδο ότι υπάρχει ε, καταγερματισμός προς ε, τις δαπάνες. Υπάρχουν ε, ε επικαλύψεις ε, στους πόρους, της ε, ικανότητας και και αυτό κοστίζει μεταξύ 25 και 100 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το 80% των ε, προκηρύξεων γίνεται σε εθνική βάση και αυτό οδηγεί ε, σε επικαλύψεις. Για να ξοδεύουμε πιο ορθά χρειάζεται ε, συνεργασία και από κοινού εργασία. Αυτό αποτελεί το νέο πρότυπο ώστε να υπάρξει προστιθεμένη αξία. Υπάρχουν κάποιοι νέοι μηχανισμοί όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα, το οποίο προσφέρει κονδύλια για έρευνα στην καινοτομία και στις τεχνολογίες. Προβλέπει 13 δισεκατομμύρια στο επόμενο πολιτισμικό πλαίσιο. Έχουμε το μηχανισμό, μηχανισμό για την ειρήνη ε, στα 10,5 δισεκατομμύρια και έχουμε και τη συνολική κινητικότητα ως ε, κομμάτι του μηχανισμού Connecting Europe που αντιστοιχεί σε 6,5 δισεκατομμύρια κατά τη διάρκεια του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου. Αυτά και άλλα μέσα θα βοηθήσουν ε, ε, γενικότερα την ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας ώστε να αυξήσουμε και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. πράγμα που αποτελεί βασικό ε, έργο όλων των πολιτικών. Σίγουρα θα ζητούν διάφορα θέματα από τους εγκεκριμένου ε, ομιλητές μας και είμαι πολύ ε, χαρούμενη που θα παρουσιάζω ο κύριος Πέντρο Σεράνο που είναι αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης υπεύθυνο για πολιτική άμυνας, για τη χρηματοδοτική πτυχή σας καλωσορίζω και σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ κύριε Σεράνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Να σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις εξελίξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές και για τις οποίες θέλουμε να έχουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χαίρομαι που ε, είναι εδώ και η κυρία Χάρντεμαν και ο κύριος ε, Πρέσα, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί στα θέματα αυτά και άλλους συναδέλφους για να δούμε πώς μπορούμε να ε, βελτιώσουμε την ασφαλή των πολιτών μας. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες τελευταία χρόνια για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να βελτιώσουμε τη, τα, την άμυνά μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα θέματα μηνάς υπερβαίνουν ε, την άμυνα. Πολλά από αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ανθρωπιστική βοήθεια και συνεργασία, ε, βελτίωση τη διακυβέρνηση και πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν κλειδί ε, για να επιδιώξουμε και την ατζέντα μα για την άμυνα. Αλλά είναι εξίσου σημαντικά αυτά που κάνουμε σε θέματα άμυνα. Όμως θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στα θέματα της άμυνας και να επενδύσουμε σε αυτήν. Είπατε κυρία Πρόεδρε ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και αυτό ισχύει και πρέπει να γίνει συλλογικά. Πρέπει να ξοδεύουμε περισσότερα αλλά και καλύτερα. Και αυτό που κάνει η σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια είναι κάτι ιδιαίτερα καινοτόμο και είναι να βοηθάει τα κράτη-μέλη να δαπανούν από κοινού σε συνεργασία πιο σωστά να επενδύουν στην ε, βιομηχανία, στην ε, τεχνολογία και στην ε, διαπιχειρηματικότητα μεταξύ κρατών μελών. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές. Είναι ένα τεράστιο θέμα και νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα μας δώσουν λεπτομέρειες, αλλά στο ευρύ πλαίσιο, αν δούμε τις προσπάθειες τα τρία κεφάλαια στο οποίο είμαστε τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο είναι η ε, ανάπτυξη στρατιωτικών ε, αμυντικών ε, δυνατοτήτων. Υπάρξουν κάποιες προσπάθειες, διερθρωμένη συνεργασία σε κάποια προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη δυνατοτήτων ώστε να μπορούμε κοινού να υποφελούμαστε το Ταμείο Άμυνας έχουμε καταφέρει να πετύχουμε πολλά με την ε, δημιουργία αυτού του που θα επιτρέψει ε, την, άμυνα, την έρευνα στην άμυνα και να φτάσουμε τα πρότυπα. Επίσης και η αξιολόγηση και αυτές ε, πτυχές έχουν κοινέ απαιτήσει. Τι πρέπει να παράγουμε από κοινού ως κρατημέλη προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν συντονιστικό μηχανισμό που θα μας ε, βοηθήσει να κατανοούμε αν κατευθυνόμαστε στη σωστή κατεύθυνση, να εντοπίσουμε ε, κοινά προγράμματα, να τα υποστηρίξουμε, να τα συμπληρώσουμε μέσω του Ταμείου Άμυνας και στο πλαίσιο του ΠΕΣΚΟ και εκτός του προγράμματος ΠΕΣΚΟ ώστε να χρηματοδοτήσουμε σχετικά προγράμματα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας αυτό και θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ και την προσφορά του Πρόεδρου της Επιτροπής που εισήκαγε για πρώτη φορά ένα νέο, ε, ένα ναι κεφάλαιο στη, στο δημοσιονομικό πλαίσιο για την άμυνα. Σε αυτά θα αναφερθεί νομίζω περισσότερο ο Σιλβάνο, οπότε θα σταματήσω εδώ και θα... Και για το Ταμείο Μήνες, αλλά και για τη στρατηγική κινητικότητα. Θα μιλήσει και για τα δύο αυτά. Όσον αφορά την κινητικότητα, είναι πολύ σημαντική για τη μετακίνηση στρατικών δυνάμεων στην Ευρώπη με αποστολές και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουμε την εδαφική αικαιρεότητα και να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις τις οποίες ήδη αντιμετωπίζουμε στην Ανατολή, ανατολικά. Αναβάθμιση των υποδομών και αντιμετώπιση ε, νομικών ε, εμποδίων που μπορεί να υπάρχουν ε, στην μετακίνηση εξοπλισμού στρατευμάτων. Υπάρχουν δομές στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και έχουμε κάνει ήδη μεγάλη πρόοδρο με τον αστυνομικό σχεδιασμό για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τι μη στρατιωτικέ ε, δυνατότητες στα κράτη-μέλη, οι οποίες τίθενται στη διάθεση τη Ευρωπαϊκής Ένωση, την ε, συνεργασία μεταξύ ε, μηχανισμών εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Θα, θα εστιάσω την προσέγγιση μου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης, στον οποίο αναφερθήκατε, ο οποίος βασίζεται στο μηχανισμό Αθήνα, Αθηνά και σε άλλους μηχανισμούς και άλλα και σε άλλα CBSD στοιχεία Έχει, έχουμε εγκαθιδρύσει λοιπόν και τον όρο άμυνα σε αυτή τη δικασία πέρα από την ασφάλεια. Το τελευταίο σημείο που έχει να κάνει με τα τρία μεγάλα κεφάλαια. Το τελευταίο είναι η συνεργασία με συνεργάτες, με εταίρους. Θέλουμε να έχουμε συνεργασία με τους εταίρους μας για να το πετύχουμε αυτό. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τον ΝΑΤΟ όλο και πιο εντατικά. Υπάρχει μια νέα κοινή διακήρυξη, η οποία υπεγράφει από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον πρόεδρο της Επιτροπής, που λαμβάνει υπόψη όλη την πρόοδο που έχουμε πετύχει τα τελευταία δύο χρόνια και που χαράζει και το δρόμο για το μέλλον αυτής της σχέσης των πυλώνα της ασφάλειας. έναν πυλώνα που έχει δύο παρακλάδια, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Το καθένα με τη δική του βαρύτητα και πολύ σχετικά και τα δύο. Ε, είναι κάτι που το πρέπει να είμαστε περήφανοι. Θα αφήσω λοιπόν τους συναδέφους ε, τον ε, Σιλβάνο να περιγράψει την αρχιτεκτονική ε, του πολιτού του μεσικού πλαισίου στο θέμα της ασφάλειας και της άμυνας και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτει αυτά τα θέματα όπως είναι ε, το Ταμείο για την Άμυνα και άλλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης. και να δούμε και τι γίνεται με το ICSP, ένα, ένα μέσο το οποίο θα τεθεί στο πλαίσιο του ICI. Η Χίλη δεν θα αναφερθεί σε αυτό, οπότε θα σταματήσω εδώ. Μπορεί να μιλήσετε πολύ, αλλά λίγα λόγια για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης, ο οποίος βασίζεται στο Μηχανισμό Αθηνά που αφορά τις ρητικές ε, αποστολές και επιχειρήσεις, το μηχανισμό ειρήνης για την Αφρική, όπου συνεργαζόμαστε με ατέρους ε, στην Αφρική υπό συγκεκριμένες συνθήκες και υπερβαίνει τους περιορισμούς που θέτουν αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα προσφέροντας πιο ισχυρή χρηματοδότηση για στρατιωτικές αποστολές μια πιο ευρεία υποστήριξη χρηματοδότηση ε, για τον εξοπλισμό των εταίρων. Αυτά είναι τα βασικά τέσσερα κεφάλαια του μηχανισμού αυτού για την ειρήνη. Όσον αφορά τις δικές μας αποστολές πλήρες του CDPS, αυτό που προτείνω είναι να ταμείο, το οποίο προβλέπει 10,5 δισεκατομμύρια για μια περίοδο 4 ετών, ώστε να χρηματοδοτήσουμε επιχειρήσεις και αποστολές ε, προσφέροντας ένα ταμείο το οποίο ήδη υπάρχει χωρίς να πρέπει να κινητοποιήσουμε νέα κονδύλια. Καλύτερη πρόσβαση, προβλεψιμότητα να γνωρίσουμε εκ των προτέρων δηλαδή τι θα, χρηματοδοτήσουμε και πιο ενισχυμένη αλληλεγγύη γιατί θα υπάρξει καταμερισμός του κόστους. Άρα θα θέλουμε να διασφαλίσουμε να υπάρχει μια πιο ισότιμη ε, συνεισφορά και χρηματοδότηση να υπάρχει ε, δίκαιο καταμερισμό του βάρου μεταξύ των κρατών μελών, Λαμβάνοντα υπόψη και τα κράτη-μέλη δεν θα, θα στείλουν αποστολέ. Ο μηχανισμό Αθηνά χρηματοδοτεί το 5 με το 10% του κόστους. Σύμφωνα με την πρόταση που έχει γίνει από την ύπατη εκπρόσωπο, θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε μέχρι το 40% αυτών των δαπανών. Αντί να έχουμε λοιπόν μια συζήτηση από τη βάση προ τα πάνω για το έχουμε μια συζήτηση από πάνω προς τη βάση, ώστε να δούμε τι θα χρηματοδοτήσουμε από κοινού και με τη βάση αυτού του ποσοστού θα αποφασίσουμε τι θα χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα. Αυτό είναι ένα καλό βήμα προς την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι η υποστήριξη ε, των επιχειρήσεων των εταίρων, όπως είναι η μηχανισμός για την ειρήνη στην Αφρική. Δεν περιοριζόμαστε εκεί στην ε, Αφρικανική Ήπειρο, αλλά την υπερβαίνουμε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, μια λύση για τη χρηματοδότηση. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση της Σομαλίας, τη Joint Farce, ε, των G5 στις χώρες του Σαχέλ, ε, για θέματα γενικά που είναι βασικά για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην Αφρική. Πρέπει να είμαστε λοιπόν σίγουροι για το τι χρηματοδοτούμε και πώς θα βοηθήσουμε άμεσα ε, και θα ενισχύσουμε την ασφάλεια της ε, Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν ένα χρηματοδοτικό μέσο που δεν ε, περιορίζεται στην Αφρική και που δεν περιορίζεται σε επιχειρήσεις που αποτελούν ε, μέρος αποκλειστικά ε, μέρος των συμπεφωνημένων ε, επιχειρήσεων με την Αφρική. Όταν έχουμε ε, με τη μετάφραση των μισών στι ε, στρατηγικέ δυνάμει τη Σομάλια, δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε το σομαλικό στρατό. Γι' αυτό, όπω λένε οι Σομαλοί, είναι ότι μα ζητάτε να αναλάβουμε αυτή τη νέα ευθύνη. Πρέπει να περάσουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο από την Αμίσον, αλλά δεν έχουμε χρηματοδοτικό μέσο αυτή τη στιγμή για να ε, στηρίξουμε τον Σομαλικό στρατό. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό και θα πρέπει να υπάρχει προστασία, παρακολούθηση, υποπτία και να δώσουμε ε, τα απαραίτητα χέγγια. Αν δεν το καταφέρουμε, τότε θα προκύψει ένα μεγάλο κενό. Το τρίο στοιχείο είναι υποστήριξη να βοηθήσουμε τον εξοπλισμό. Υπάρχουν περιορισμοί με το τρέχον χρηματοδοτικό μέσο και εντός του Μηχανισμού για την Ειρήνη στην Αφρική. Π.χ. στην Κεντρική Αφρική δεν είχαμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε ε, όπλα πράγμα για την Κεντρική Δημοκρατία της Αφρικής που δημιούργησε προβλήματα στην ε, ενίσχυση της ασφάλειας. Άρα εδώ χρειάζεται ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλοί έλεγχοι, να τεθούν σε ισχύ πολυελεκτικοί μηχανισμοί ώστε να διασφαλιστούν τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό, άμα δεν προβούμε σε αυτό το ούτε δεν θα βοηθήσουμε ούτε τη δημοκρατία ούτε τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία λοιπόν αυτού του νέου χρηματοδοτικού μέσου. Είναι αρκετά καινοτόμο. Για πρώτη φορά έχουμε ένα άρθρο θήκη που επιτρέπει στην υπάντη εκπρόσωπο να κάνει προτάσει με την υποστήριξη τη Επιτροπή. Να ευχαριστήσω και πάλι του συναδέλφου από την Επιτροπή. Η Χίλντε έχει εργαστεί πολύ σκληρά για να μας δώσει όλες τις εγγύσεις ενός αποδοτικού μέσου, ενός αξιόπιστου μέσου και θα παραχωρηθεί η δημοσιονομική διαχείριση στο FBI μετά από προτάσεις που θα γίνουν από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Οι αποφάσει για το πώ θα γίνει η διαχείριση αυτή από τα κράτη-μέλη είναι έγκυτες στα ίδια τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα αντιπροσωπεύονται και στη Διαχειριστική Επιτροπή και σε σχέση με τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές και τις πολιτικές. θα απαιτείται ομοφωνία για τα πρώτα κεφάλαια, ενώ για τα άλλα δύο κεφάλαια θα απαιτείται η ενισχυμένη πλειοψηφία στις ψηφοφορίες και η οικονομική διαχείριση θα είναι στα χέρια της FBI. Ο δημοσιονομικός κανονισμός θα είναι ειδικό για την περίπτωση, όπως έχουμε και για το EDF, θα υπάρξει και ένας μηχανισμός εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, τον οποίο θα ελέγχει το ελεγκτικό συνέδριο. θα είναι ανοιχτή στην Αφρική αυτή η δυνατότητα, το μέσο αυτό είναι βασικό στόχος για τη χρήση του μηχανισμού η Αφρική και αναφέρεται αυτό και στο προήμιο. 10,5 δις δεν έρχονται από το πουθενά. Υπάρχει σαφής υπολογισμός με βάση τις εμπειρίες τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα. Ελπίζω ότι αυτό θα ανήκει και στη συζήτηση για το ε, πολιετές δημοσιονομικό στο μέλλον. Είναι μεν εκτός προϋπολογισμού, αλλά έχει σχέση με το σύνολο των καταβολών των χωρών προς τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ε, μακρηγόρησα, ζητώ συγγνώμη για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να είμαι εδώ με τους εκλεκτούς συναδέλφους μου. Είμαστε στην υπηρεσία σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και για την λεπτομερέστατη παρουσίαση Απαντήσατε και σε πολλές πιθανώς ερωτήσεις που θα τεθούν. Ο επόμενος ομιλητής ε, είναι προσωρινός διευθυντής ε, της ε, Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι αυτός από τον οποίο θα περάσουν και τα χρήματα για τα οποία επίσης συζητήσαμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας μεταφέρω τις δράσεις της Επιτροπής στον τομέα της άμυνας και τι προτείνουμε για το επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό. Θα περιοριστώ στα θέματα τα δημοσιονομικά και πώς αυτό εντάσσεται και στο ισχύον ε, ε, δημοσιονομικό πολιετές. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Περιλαμβάνεται στην πρόταση και για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το τι υπάρχει ήδη καταρχάς, υπάρχουν παρασκευαστικές δράσεις στον τομέα της έρευνας για την άμυνα από το 2007 μέχρι το 2019. Ξέρετε ότι δεν μιλάμε μόνο για θέματα άμυνας, αλλά υπάρχουν και κάποια επιμέρους προβλήματα πολυδιάσπασης τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τις δαπάνες αυτές και η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι να δώσουμε κίνητρα για τη βελτίωση της συνεργασίας και την βελτίωση της ε, αποτελεσματικότητας των χρημάτων τα οποία δαπανώνται στον τομέα της άμυνας. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχετε 13 συστήματα όπλων ενώ έχετε 178 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εκ τούτου λοιπόν η αποτελεσματικότητα των δαπανών επηρεάζεται αρνητικά σε σχέση με τις προπαρασκευαστικές δράσεις έχουμε πετύχει κάποια αποτελέσματα έχουν υπογραφεί οι πρώτες συμβάσεις έχουν ξεκινήσει σε σχέση με τα drones και τα αντίστοιχα υποβρύχια σκάφη και θα ήθελα εδώ να χαιρετήσω τις προσπάθειες και την επικοδομητική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πρόγραμμα έρευνας για τον τομέα της άμυνας. Αποφασίστηκε πρόσφατα αποφασίστηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και σε δημοσιονομικά επίπεδο υπάρχουν 500 εκατομμύρια που θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό από το 19, για το 19 και το 20 και αυτό θα δημιουργήσει κίνητρα για τα κράτη-μέλη να πάρουν μέρος στην προσπάθεια και ελπίζεται δύο δις να προέλθουν από τα κράτη-μέλη μεμονωμένα ε, σε κοινούς στόχους, σε κοινά προγράμματα στην αναπτυξιακή αρχική φάση έτσι ώστε να πετύχουμε την επιθυμητή αποτελεσματικότητα. Ε, μετά έχουμε την βάση θα έλεγα της πρότασης για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό. Εδώ η άμυνα αναλαμβάνει αν θέλετε και μία νέα διάσταση και περιλαμβάνει πολλές νέες προτεραιότητες οι οποίες ε, χαρακτηρίζουν την πολιτική της Αφρικής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί διαφθρωτικά στην αρχιτεκτονική του προϋπολογισμού Υπάρχει ένα συγκεκριμένος τίτλο στον προϋπολογισμό πλέον για την άμυνα και την ασφάλεια. Αυτό θα φαίνεται και στο πολιετές δημοσιονομικό και στα πλαίσια αυτή της συγκεκριμένης δαπάνης θα υπάρχει ένα ξεχωριστό σύνολο γραμμών για την άμυνα. Εδώ θα έχουμε δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ένα θα παραπέμπει άμεσα στα θέματα της έρευνας και σχετικά με τα 4,1 δις και μετά έχουμε τα υπόλοιπα τα οποία σχεδόν 19 που αναφέρεται στις επιχειρησιακές δυνατότητες. Σε σχέση με τους στόχους τους οποίους έχουμε είναι προφανές η προσπάθεια ανάπτυξης μιας κάποιας στρατηγικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουμε να κάνουμε με τις δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε να κάνουμε με θέματα προώθησης τεχνολογικής καινοτομίας και έρευνας. Έχουμε να κάνουμε με θέματα ενίσχυσης συνεργειών με τους υπόλοιπους εταίρους στον τομέα της άμυνας και επίσης έχουμε να κάνουμε με μορφές ενίσχυσης της συνεργασίας και των συνεργειών και με τις υπόλοιπες πολιτικές, όχι μόνο ασφάλεια, αλλά ασφάλεια γενικότερα και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνεκτικότητα. Σε σχέση με τις συνέργειες οι οποίες προβλέπονται θα υπάρχει και σε σχέση με άλλες πολιτικές όπως η έρευνα φυσικά θα υπάρξει διασταυρούμενη γονιμοποίηση αν θέλετε ανάμεσα στην έρευνα που γίνεται για πολιτικά, για μη στρατιωτικά ε, πεδία και από την άλλη για στρατιωτικούς ε, λόγους. Ξέρετε ότι το παράδειγμα το κλασικό είναι το διαδίκτυο. Το ίντερνετ δημιουργήθηκε σαν στρατιωτικό ε, μέσο, αλλά παρόλα αυτά επεξετάθηκε στον τομέα των μη στρατιωτικών. Θα υπάρχουν επίσης συνέργειες και με τα διαστημικά προγράμματα σε σχέση κυρίως με τα GPS και ταυτόχρονα θα υπάρξουν και συνέργειες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σχετικά με την πρόταση που έχει γίνει η ψηφιακή Ευρώπη, το Digital Europe ε, και το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολιετούς δημοσιονομικού. Θα υπάρξουν επίσης συνέργειες και σε άλλα προγράμματα όπως ε, η έρευνα στον θαλάσσιο ε, τομέα και η κοινή ατζέντα στρατιωτικής και μη στρατιωτικής χρήσης. Υπάρχουν συνολικά λοιπόν 19,5 δίσες συνολικά για την κάλυψη των αναγκών αυτού του συνόλου των αμυντικών θέσεων στον προϋπολογισμό για, τα επόμενα, για το επόμενο δημοσι... Ε, πολιετές δημοσιονομικό συν το 5,1 δις τα οποία θα χρηματοδοτηθούν εκτός προϋπολογισμού για το European Peace Facility, για το ειρηνευτικό μέσο Υπάρχουν περιορισμοί για το τι μπορεί να χρηματοδοτήσει ο προϋπολογισμός αυτός, περιλαμβάνονται στην ίδια συνθήκη, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ο προϋπολογισμός αποκλειστικά στρατιωτικής και αμυντικής φύσης. Συνεπώς υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το νέο προϋπολογισμό είδαμε την δυνατότητες βελτίωσης των επιχειρησιακών ικανοτήτων μπορεί να υπάρξει αλλά κάποιες δράσεις αυστηρά στρατιωτικού χαρακτήρα που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και στα οποία αναφέρθηκε ο προλαλής σας, μπορεί να καλυφθούν έξω του από τον προϋπολογισμό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιετές δημοσιονομικό και η πρόταση του υπάτου εκπροσώπου για την Ευρωπαϊκή για το Ευρωπαϊκό Ειρηνευτικό Μέσο θα πρέπει να ειδωθούν από κοινού με συνδυαστικό τρόπο. Ξέρω ότι ο πρόεδρος Αρτουή δεν είναι οπαδός της χρηματοδότησης μέσων εκτός προϋπολογισμού από άλλες πηγές ενώ. αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβουμε υπόψη μας το τι ε, προβλέπει το διακανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμεθα να λειτουργήσουμε δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε και τελικά εξαρτάται από αυτό και η αποδοτικότητα των, της χρήσης των πόρων, των διαθέσιμων πόρων. Σε σχέση με την ένταση της προώθησης της συνεργασίας σε νέους τομείς, στην έρευνα και στην ανάπτυξη επιχειρησιακών ικανοτήτων, ε, η στήριξη του δημοσιονομικού αν θέλετε πλαισίου θα ε, καθορίσει και ε, τις δυνατότητες που θα έχουμε σε τομείς όπως η έρευνα, στον τομέα της δημιουργίας πρωτοτύπων θα υπάρχει η δυνατότητα πριν περάσουμε στη σχεδίαση του πρωτοτύπου μέχρι 100% και όταν φτάσουμε στην φάση κατασκευής του πρωτοτύπου τότε θα πέσει στο 20% του συνολικού κόστους και μετά από την φάση του πρωτοτύπου μπορεί να ξανανεύει πάλι στο 80% σαν παράδειγμα για τις διαδικασίες πιστοποίησης. Α, επιπλέον για να υπάρξει και μια κάποια ενθάρρυνση για την κοινή προσπάθεια προβλέπονται διάφορα μπόνους στα πλαίσια της διαφθρωτικής συνεργασίας υπάρχει η δυνατότητα σαν παράδειγμα 10% μπόνους επιπλέον των προηγούμενων ποσών και το ίδιο ισχύει και για προγράμματα τα οποία προωθούν την διασυνοριακή συνεργασία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω ενθάρρυνση δημιουργίας βιομηχανικών δομών διασυνοριακών. να μου επιτρέψετε να πω λίγα πράγματα τώρα. για θέματα εφαρμογής των προγραμμάτων τα οποία καλούμεθα να χρηματοδοτήσουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσει εδώ. Πρέπει να υπάρχουν ε, τρεις τουλάχιστον χώρες μέλη για να διασφαλίζεται ο διασύνοραϊκός χαρακτήρας ε, οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν έδρα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ελέγχονται από εταιρείε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχική διαχείριση και ο έλεγχος διαχείρισης να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα θέματα τα εφαρμοστικά να οργανώνονται με βάση τα ετήσια και πολυετή ε, προγράμματα εργασίας. Όπως είπε και ο κ. Σεράνο, ε, τα προγράμματα θα αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Να προσθέσω τώρα κάποια σημεία σχετικά με την στρατιωτική κινητικότητα. Μιλάμε για 6,5 δις τα οποία προβλέπονται επιπλέον των 13 δις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας Συνολικά φτάνουμε στα 20 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια του επομένου δημοσιονομικού. Εδώ η τεκμηρίωση αν θέλετε γίνεται ως εξής. Δημιουργία μόχλευσης, δημιουργία συνεργειών για προγράμματα υποδομών τα οποία είναι λεγόμενη διπλής ειδητής χρήσης και για πολιτικούς λόγους, για λόγους μη στρατιωτικούς να είναι προγράμματα τα οποία θα διευκολύνουν όμως και την μετακίνηση στρατευμάτων ή μετακίνηση στρατιωτικών εξοπλισμών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να διευκολύνονται ε, στρατιωτικά γυμνάσια, δοκιμές αλλά και ε, όταν υπάρχουν κατεπίγουσες καταστάσεις να διασφαλίζεται η γρήγορη αντίδραση σε επίπεδο δημοσιονομικό. Αυτά όλα συνδέονται επίσης και με τα λεγόμενα TEN και ταυτόχρονα σε σχέση με τη νομική βάση και τις δυνατότητες χρηματοδότησης εντάσσονται και στο μέσο Connecting Europe, στον τομέα, ε, στον κλάδο των μεταφορών. Συνεπώς λοιπόν είναι διασφαλισμένη η νομική βάση. Ε, δεν θα μακρηγορήσω άλλο, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις σε ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια ε, θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις. Έχουμε και τρίτη ομιλήτρια όμως, που είναι η κυρία Χίλντα Χάρντεμαν, επικεφαλής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Μέσα Εξωτερικής Συνεργασίας και ακριβώς όταν έχουμε χρηματοδότηση εξωτερικών δράσεων όπως είναι αποστολές ΕΠΑ είστε εσείς αρμόδια. Παρακαλώ κυρία Χάρτμαν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι ενώπιον σας για να ενισφέρω και εγώ στη συζήτηση αυτή. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στην ε, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης ε, στο γενικότερο πλαίσιο της ΕΠΑ και να συμπληρώσω ε, ορισμένα ε, από τα όσα είπε ο προλαλής σας κύριο Σερανό από τη σκοπιά της διοίκησης και διαχείρισης. Η υπηρεσία της οποίας συγούμε εξασφαλίζει ε, την οικονομική διαχείριση των πολιτικών, μη στρατιωτικών μέσων για την πρόληψη των σειράξεων, τη σταθερότητα και την ειρήνη. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ιστορικό υγιούς ε, δημοσιονομικής διαχείρισης αλλά και δημιουργικότητας ε, και αποδοτικότητας. Μέσω ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού έχουμε διάφορες δυνατότητες. Έχουμε το μηχανισμό για τη σταθερότητα και την ειρήνη, για ταχεία απόκριση σε περιπτώσεις κρίσεων και για πρόληψη σειράξεων. Μετά από πάρα πολύ στενή συνεργασία που είχαμε πέρσι με το Ευρωπαϊκό ε, κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καταλήξαμε σε ένα μέσο που μπορούμε πλέον να συνεργαζόμαστε και με στρατιωτικούς, ιδιαίτερα για τη δημιουργία επιχειρησιακών ε, ικανοτήτων, ε, το λεγόμενο CPSD. Τα γνωρίζετε αυτά τα θέματα και τις ειδικέ συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός. Πρώτον, αν υπάρχει σοβαρή απειλή ε, προς ε, θεσμούς ή σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και των θεμελιωδών ελευθεριών. Δεύτερον, όταν κάποιοι στρατιωτικοί φορεί είναι οι μόνοι που μπορούν να επιφορτιστούν με ένα συγκεκριμένο έργο. Και τρίτον, όταν υπάρχει και συνένεση Ευρωπαϊκή Ένωση και του εν λόγω κράτου ότι χρειάζεται οπωσδήποτε επέμβαση των στρατιωτικών δυνάμεων για να εκτελεστούν αυτά τα έργα. Το πρώτο έργο ή τα πρώτα μάλλον τώρα εκτελούνται αυτό το καιρό και στο μέλλον η ταχεία αντίδραση θα πρέπει να παραμείνει βασικό στοιχείο του πλαισίου μετά το 2020 και της μεταρρύθμισης του νέου πυλώνα στην, ε, στα διάφορα μέσα για τη διεθνή συνεργασία, την ανάπτυξη και την πολιτική γειτονίας. Πέρα από αυτές τις δράσεις ταχείας αντίδρασης υπάρχει και ένα νέο και ένα άλλο σκέλο που είναι η υποστήριξη των ε, πολιτικών μη στρατιωτικών αποστολών ΕΠΑ μπορεί να αναπτύσσεται ταχύτητα, ταχύτατα και να ε, δρά ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Αυτές οι αποστολές ε, λειτουργούν σε δύσκολα περιβάλλοντα και ε, σε αισθήσει κρίσης. Η υπηρεσία μας έχει την εποπτεία επισκόπηση και την οικονομική διαχείριση. Οι αποστολές αυτές έχουν μεγάλη ζήτηση καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πρωταγωνιστή στη διεθνή διαχείριση, πολιτική διαχείριση των κρίσεων. Ε, και Χαιρόμαστε για την υποστήριξη ε, από την Επιτροπή σας σήμερα το πρωί για να μπορούμε να εργαστούμε σε αυτό το πεδίο εφαρμογής. Ακριβώς επειδή έχει μια ιδιαιτερότητα ο προπολογισμό αυτό για τη χρηματοδότηση πολιτικών αποστολών, θα παραμείνει αυτό χωριστό εργαλείο και στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τουλάχιστον αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ θα πρότεινα να επεκταθεί ε, και να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Αλλά, γιατί εδώ έρχεται και ένα αλλά, όσο πολύτιμα και να είναι αυτά τα μέσα εντός του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να παραμείνουν και να ενισχυθούν έτσι περαιτέρω οι δραστηριότητε και τα μέσα στο επόμενο PDP. Υπολείπονται όμω για του λόγου που εξήγησε ο κύριο Πρέζα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δράσει με σαφή ε, στρατιωτική ή αμυντική διάσταση. Αυτό είναι ένα κομμάτι της εικόνας που θα πρέπει να συμπληρωθεί και από ένα δεύτερο, δηλαδή μέσα εκτό προπολογισμού που μπορούν να χρηματοδοτήσουν στρατιωτικές ή αμυντικέ διαστάσεις. Ε, και εδώ ε, έχουμε το μέσο, το μηχανισμό ε, για την σταθερότητα και την ειρήνη που περιέγραψε ο κύριος Σεράνο. Θα πρέπει εμεί να διαδραματίσουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ότι εκπρόσωπο είπε ότι θα μας επιφορτήσει και με την οικονομική διαχείριση ε, αυτής ε, του, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης. Είναι σαφής η λογική. Από τη μια δική μας υπηρεσία υπάγεται ε, στην κυρία Μογκερίνη και από την άλλη έχει και ρόλο ήδη οικονομικής διαχείρισης των άλλων μέσων που σας ανέφερα προηγουμένως. Οπότε είναι κατάλληλη και έχει και την ιδεώδη εμπειρία για να φορτιστεί με αυτό το έργο. Θα συνεργαστούμε ε, και με άλλα ε, εργαλεία εξωτερικής δράσης στην προσπάθεια αυτή, τα οποία ήδη διαχειριζόμαστε για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ένα από τα βασικά σχέδια του μηχανισμού αυτού είναι η δυνατότητα ενίσχυσης για επιχειρησιακές ικανότητες σε στρατιωτικούς φορείς, ε, γιατί χρειάζεται πολύ, πολλές φορές υποστήριξη όπου δεν επαρκούν ε, ή δεν βρίσκουν εφαρμογή τα στοιχεία που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό ε, Υπολογισμό που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν στρατιωτικές ή αμυντικές δράσεις. Λοιπόν, για να κλείσω οι νέες δομές που προτείνονται στο επόμενο PDP και οι ε, δομές για την ειρήνη ε, θα συμβαδίζουν και θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερες συνέργειες μέσα στις υπηρεσίες μας για να μπορούμε ε, με τρόπο αποτελεσματικό και γρήγορο να ανταποκρινόμαστε στις προτεραιότητες της Ένωσης για την ασφάλεια και τη σταθερότητα είναι στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστολή της να εξασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα και οι στρατηγικές πολιτικές επιλογές αφορούν και τη δική μας εργαλειοθήκη. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία ακριβώς την εργαλειοθήκη μας για να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση απολύτω και πλήρως το ρόλο της για την ασφάλεια των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές μας και με μεγάλη χαρά θα ξαναδώσω την Προεδρία στον κύριο Ορτουή. Χαχα. Ήσασταν ε, ε, πραγματικά θαυμάσια πρόεδρος. Ευχαριστώ και πάλι και τους τρεις ομιλητές. Χαιρετίζω την εφευρετικότητα του συστήματος. Θα με παρεξηγήσει ο κύριος Πρέζα. Ξέρετε ότι εγώ είμαι υπέρ του ενιαίου χαρακτήρα του προπολογισμού. Γιατί θα πρέπει ο προϋπολογισμός να μιλάει και στους Ευρωπαίους πολίτες. Όταν τους λέμε ότι ε, ε, ασχολούμαστε με την ε, άμυνα, αλλά όχι και ακριβώς, γιατί έχουμε ξεχωριστό κεφάλαιο, θα πρέπει η Ευρώπη με σαφήνεια και με ενιαία μορφή να προβάλλεται στους Ευρωπαίους πολίτες. Η κυρία Τομάζη, σε πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λοιπόν τους ε, προηγούμενους ομιλητές. Καταρχάς θα ήθελα να... Bien sûr. Euh, να χαιρετήσω την κυρία Μούντι για την επιστροφή της. Εγώ δεν υποτιμώ καθόλου την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Δεν θα μιλήσω όμως για τέτοιου είδους θέματα. Είμαστε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι πάντα ήμουν απεπισμένος για την αξία της Ευρωπαϊκής Άμυνας, ιδιαίτερα στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο, αυτή η πεποίθησή μου ενισχύεται. Όμως, ε, εμείς έχουμε να ασχοληθούμε για θέματα που άρτονται της Επιτροπής μας. Ξεχάσατε την ψήφο του Κοινοβουλίου σε σχέση με τη σύνθεση. Καταρχάς, για το θέμα του εκτός προϋπολογισμού χρηματοδοτούμενο. Όπως είπε ο πρόεδρος Σαρτιουή, ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, εντελώς υποκριτική Υποτίθεται ότι δεν μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, οπότε παραβιάζουμε τις συνθήκες και φτιάχνουμε ένα εξωτερικό προϋπολογισμό. Γιατί το θέμα τίθεται ως εξή ή πράγματι τα κράτη-μέλη είναι πεπισμένα και να αλλάξουν τον κανόνα, αλλά όχι να παραβιάζουν τη συνθήκη. Η αποτελεσματικότητα δεν πρέπει να αμφισβητεί την ειλικρίνεια. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ λοιπόν και θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο Τρίκ. Τώρα, τα έσοδα. Πράγματι, συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Το θέμα είναι βέβαια με τι χρήματα. Με τι χρήματα θα γίνει. Το κοινοβούλιο έχει κουραστεί λιγάκι και έχει εκνευριστεί γιατί βλέπει το Συμβουλίο να ανακοινώνει όλο και περισσότερες δαπάνες χωρίς ποτέ να θέτει το θέμα των πόρων, λέγοντας ότι καλά δεν πειράζει, θα κάνουμε περικοπές στον υπάρχοντα προϋπολογισμό, ανεξάρτητα πού και πώς θα τις κάνουμε, γιατί βασικά έχουμε νέες προτεραιότητες κάθε φορά. Οπότε βρισκόμαστε σε μια εντελώς παράλογη κατάσταση, με ένα πολιετές δημοσιονομικό το οποίο δεν δουλεύει λόγω των συνεχών περικοπών. Προσέξτε για την άμυνα, γιατί αυτό μπορείτε να πάθετε και εσείς αύριο. Μια νέα προτεραιότητα μπορεί να υπάρξει, οπότε θα χάσετε εσείς τα λεφτά σας. Συνεπώ λοιπόν δεν θα είναι επαρκή η χρηματοδότηση. Ανησυχούμε λοιπόν όταν βλέπουμε ότι ένας προϋπολογισμός, ο οποίος ήταν προϋπολογισμός κυρίως αλληλεγγύης, ταχύτατα, να γίνεται προϋπολογισμός αμυντικός, αν και δεν είμαι εναντίον ενός αμυντικού προϋπολογισμού. Να διευκρινίσω και το επιπλέον πρόβλημα το οποίο εμείς περιλαμβάνουμε στην θέση την οποία πήραμε πρόσφατα και περιμένουμε ακόμα την απάντηση ότι δεν έχουμε προβλήματα με τις νέες προτεραιότητες με την προϋπόθεση ότι θα αυξηθεί και ο προϋπολογισμός. Αυτή είναι η πρόταση την οποία είχαμε κάνει. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια πρώτη ψήφος για τα προπαρασκευαστικά. Και αυτό το οποίο σας είπα μόλις επικυρώθηκε. Από τη μία χρησιμοποιήθηκαν τα περιθώρια της ε, ευελιξίας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλα χρήματα εκεί, οπότε στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό θα πρέπει να πείτε στους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο, στους φίλους σας στο Συμβούλιο, ότι το πράγμα δεν πάει έτσι. Οπότε ή θα συνεχίσουν τις περικοπές, οπότε θα τους αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο, ε, δεν θα υπονομεύσουν πια όπως κάνουν σήμερα τις πολιτικές συνοχής και τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές αλληλεγγύης. Έχουμε ένα πρόβλημα λοιπόν πόρων, θα είμαστε σκληροί, δεν είναι όπως έλεγε ο τίτλος του παλιού ντοκιμαντέρ στο βάθος που έρχεται από μακριά φαίνεται η, ε, η καταιγίδα, δυστυχώς θα την προλάβουμε εμείς από δική μας πλευρά και υπάρχει και ένα επιμέρος τιμίο, ε, μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια. Ένας από εσά δεν ξέρω ποιος, δεν πρόσεξα το όνομα, ίσως ο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρίνησε ότι η πρόταση είχε γίνει με βάση την δυνατότητα δύο κρατών, ενώ εμείς είχαμε προτείνει τρία κράτη για την ελάχιστη αποδεκτή πρόταση. Ε, Διαρωτώ με λοιπόν τι στο καλό κάνει ένας νομοθέτης εδώ και θα ήθελα τη θέση σας γύρω από αυτό. Καλώ, τελειώσατε κύριε Τωμά. Α, προς το παρόν. Μάλιστα. Ο συνάδελφος Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αλλά θα τα πω στα αγγλικά. Θα ξεκινήσω με γενικές παρατηρήσεις. Υπάρχει πλέον μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ της ε, πολιτικής συνοχής μεταξύ των κρατών μελών, συνοχή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και την ασφαλεία και την άμυνα. Γιατί η ασφάλεια μπορεί να αποδειχθεί ένα μεγάλο εφόδιο την ε, συνοχή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, υποστηρίζω την ε, ιδέα του να ξεκινήσουμε την οικοδόμηση μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Τα νούμερα δεν είναι τόσο εντυπωσιακά. Μπορεί το 2017 να είχαμε λιγότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ συν ε, το σωρευτικό παράγοντα Παρ' όλα αυτά όμως οι δαπάνες σε εθνικό επίπεδο είναι ελάχιστες. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να την τρέξουμε ε, αυτή την πολιτική παράλληλα με το νέο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή και την Επιτροπή Εξωτερική Δράση πώ πώς προσδιορίζετε τις βασικούς τομείς, στους οποίους πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τα νέα προγράμματα άμυνας, γιατί με τις άποψεις ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο ε, ο κυβερνοχώρος όπου τα κράτη-μέλη που ε, θα πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα, να συγκεντρώσουν πόρους και ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο ώστε να έχουμε τις δυνατότητες να αμυνθούμε γιατί τώρα δεν υπάρχει ένα κράτος μέλος που να μπορεί να το πράξει αυτό με ίδιους με δικούς του πόρους. Ακόμα και τα πιο καλά εξοπλισμένα κράτη-μέλη όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία ή το Βασίλειο δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν αυτό μόνα τους. Το δεύτερο έχει μεγάλη αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να επενδύσουμε σε τομεί όπου υπάρχουν ε, εντυπωσιακέ νέες εξελίξεις όπως είναι τα drone, τα laser και θα πρέπει η Ευρώπη με την ε, τεχνογνωσία να κάνει τη διαφορά και να ε, συμπληρώσει το κενό στο να δώσει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα. Το άλλο έχει να κάνει με τη στρατηγική κινητικότητα Πώς θα γίνει σωστή εφαρμογή. Υπάρχουν, ε, υπάρχει διάσπαση στο Κοινοβούλιο ως προς το αν θα μεταφερθούν τα 10 δισεκατομμύρια στο μηχανισμό Connecting Europe ή θα είναι λιγότερο από 10 δισεκατομμύρια. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρα κριτήρια για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στο μηχανισμό Connecting Europe και παράλληλα να έχουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό γιατί χρειάζεται να επενδύσουμε στην πρώτη φάση κινητικότητας που είναι και η πιο απαραίτητη. Και αναφέρομαι και θα από αυτό που είπε η καγκελάριος Μέρκερ, χρειάζεται να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας στην άμυνα στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης όπου υπάρχει μία άμεση ε, απειλή για την ασφαλειά μας από τη Ρωσία. Γι' αυτό αυτό ο στρατηγικό σχεδιασμός με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη είναι σημαντικός γιατί αυτή είναι μια στρατηγική άσκηση. Δεν μπορούμε να την κάνουμε βραχυπρόθεσμα προσπαθώντα να γεμίσουμε μικρά κενά. Θα πρέπει να είναι συνεκτική, να είναι ε, ένας ενιαίος σχεδιασμός που θα μας επιτρέψει ω Ήπειρο να έχουμε τη ε, δυνατότητα να μεταφέρουμε εξοπλιστικό μηχανισμό στρατεύματα όταν είναι απαραίτητο. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω την εκπρόσωπο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης αν έχουν σκοπό να, να κάνουν προσαρμογές σε πρωτόκολλα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με μεταφορές εξοπλισμού, έχει να κάνει και με προσωπικό. Δεν μπορείτε να πείτε στον κύριο είναι να κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ και μετά θα δούμε πώς θα τοποθετήσουμε τα στρατεύματά μας πρέπει να κάνουμε ε, προσεκτικό σχεδιασμό, να προετοιμάσουμε τα πρωτόκολλα, ώστε να μπορούμε να τα αναπτύξουμε με τρόπο ταχύ. Ταυτόχρονα ενθαρρύνω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αποτρέψουν την διάσπαση απόψεων να αποφευχθούν αυτές οι ανούσιες ε, ε διαφωνίες που απειλούν ε, την αλληλεγγύη και την ενότητα. Γιατί η πολιτική άμυνας μπορεί να αποβεί σε όφελος μιας ε, ένωσης. Άλλος, ο Τάραντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι όπλο διτής χρήσης εδώ, γιατί εκπροσωπώ την κυρία Βαλέρο από την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και είμαι και από την Επιτροπή Προϋπολογισμό για να μειώνουμε τις δαπάνες. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Κυκλοφόρησε ένα έγγραφο για τη σημερινή συνεδρίαση που κάνει αναφορά στο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες, το 2% του ΟΕΠ. Και υπάρχει το επιχείρημα ότι το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και άλλα μέσα που έχουμε θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε και να καλύψουμε το στόχο αυτό του ΝΑΤΟ. Για χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, βλέπετε Σουηδία, Αυστρία, Ιρλανδία και Φιλανδία, αυτό από νομικής απόψεως μπορεί να αποδειχθεί προβληματικό. Δηλαδή να συνεισφέρει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, στις αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών για σκοπούς του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, η συλλογική άμυνα της επικράτειάς μας μέχρι σήμερα και θα δούμε προσεχώς τι θα πει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, είναι από τα βασικά ε, καθήκοντα του ΝΑΤΟ αλλά δεν αναφέρεται στη συνθήκη τη δική μας, αλλά τα νέα μέσα του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου επικεντρώνονται πάρα πολύ σε αυτά. Πώς όμως αυτά που αποφασίζετε συνάδουν με τα όσα λέει η συνθήκη για τα στρατιωτικά. Το δεύτερο, το θέμα των στρατιωτικών μεταφορών εξετάζουμε μια πρόταση να πάρουμε χρήματα από τη διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη, ΣΕΦ, για να τα αφιερώσουμε εκεί. Για πολλούς αυτό σημαίνει ότι θα φύγουν άρματα από τη Δύση να πάνε ε, στην Ανατολή, ξέρω εγώ, σιδηροδρομικός κτλ. Υπάρχει όμως στη Βαλτική ένα πολύ προβληματικό σχέδιο. Rail Baltica. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα γίνει αυτός ο σιδηρόδρομος για να αναπτύσσονται στρατηγικές, στρατιωτικές δυνατότητες στη Βαλτική. Πάνε 110 χρόνια από τότε που τα τεθροκισμένα τρένα έκαναν τη διαφορά στα πεδία των μαχών. Εκεί έχουμε γυρίσει. Δηλαδή θα πάρετε όλα αυτά τα χρήματα από τις χώρες της Βαλτικής για, να χαράξετε αυτή τη συνδρομική γραμμή. Γιατί δεν θα έρχονται από εκεί τα κινέζικα εμπορεύματα, ούτε τα θωρακισμένα τρένα. Και το, εδώ σταματώ τις σκέψεις της κυρίας Βαλέρο. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη ένα στον άλλο και όχι δυσπιστία και καχυποψία. Και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε λεπτό του ευρώ που δαπανούμε εκεί πιάνει τόπο. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι δαπανούμε για την άμυνα. Και να μην χτίζουμε και άλλα κτίρια από όλα ρίσπαξ στις Βρυξέλλες. όπου εδώ πέρα έρχονται διάφοροι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν ξέρω να κάνουν τίποτα, ή δεν είναι ικανοί να κάνουν τίποτα για την άμυνα. Σταματώ εδώ. Merci, Ευχαριστώ κύριε Τάραντ. Άλλο. Δεν ζητεί κανεί άλλο συνάδελφο τώρα λόγο. Θα ήθελα καταρχά εγώ να καλωσορίσω το παιδαγωγικό χαρακτήρα του εγγράφου που εκπώνησε η Διεύθυνση Προϋπολογισμών, έτσι δεν είναι, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ωραία αυτή η απεικόνηση των διαφόρων οπλικών συστημάτων. 178 στην Ευρώπη και 30 μόλις στις Ηνωμένες Πολιτείες. 17 τύποι αρμάτων μάχης, ένα μόνο έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, φρεγάτες και αντιτορπιλικά, 29 στην Ευρώπη, 4 ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Καταδιοκτικά μαχητικά αεροσκάφη, 20 στην Ευρώπη τύποι, 6 στις Ηνωμένε Πολιτείες. Οι Ευρωπαίοι όμω ακρεφνεί υποστηρικτέ τη Ευρωπαϊκή Άμυνας, πάνε και αγοράζουν όπλα από τι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούσαμε να δούμε εδώ τι τύποι οπλικών συστημάτων είναι Ευρωπαϊκή κατασκευή και ποια ε, έχουμε αγοράσει shelf, έτοιμα δηλαδή από τι Ηνωμένες Πολιτείες ή απαλού. Για να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πνεύμα, γιατί καλό είναι να έχουμε μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Αλλά αν τα μέλη της ΠΕΣΚΟ εξακολουθούν να ψωνίζουν πυράβλους Patriot και, και τέτοια ε, ελικόπτερα ή ε, καταδιοκτικά άλλο, καλό θα ήταν να τα συζητήσουμε. το Το δεύτερο ερώτημα αφορά την ΠΕΣΚΟ. Τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Υπάρχει χωριστό ειδικό προπολογισμό για αυτή και πώ λειτουργεί, αν δεν έχει ειδικό προπολογισμό. Είναι απλώς μια χαλαρή σχέση συνεργασίας, η δημοσιονομική έκφραση έχει και ποια είναι αυτή. Και τρίτη παρατηρήση για τη συνθήκη. Διότι εμείς εδώ εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε τώρα λοιπόν μια άσκηση ε, ε, στο περιθώριο των συνθήκων. Ενώ υπάρχει μια ολόκληρη σχολή σκέψης στην Ευρώπη, ε, που θα ήταν υπέρ ε, ε, μιας ευρωπαϊκής άμυνας κανονικής. Μήπως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση των συνθήκων. Καλά είναι να προσπαθεί να κερδίζει έδαφος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα ισχυρότερο και θα πρέπει να εκφράζεται και στην πολιτική συζήτηση. Είναι θέμα δημοκρατικής νομιμότητας αυτό και νομιμοποίησης. Καλά, δεν θα επανέλθω στην ανάγκη της ενότητας του προεπλογισμού καταλάβαμε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι αστερισμός ε, μέσων διευκολύνσεων, μηχανισμών, ταμείων, ε, καταπιστευμάτων και πάει λέγοντα. Αλλά ε, αντικειμενικά οι πολίτες δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Δηλαδή τίθεται ένα θέμα δημοκρατικότητας. Και αν θέλουμε να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή άμυνα δεν μπορούμε να πούμε ότι κοιτάξτε οι εθνικές αμυντικές δαπάνες δεν είναι αποτελεσματικές και καλό θα ήταν ε, αυτές οι πιστώσεις που είναι πολύ σατελές φορές στα κράτη-μέλη να τεθούν ε, στη διάθεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και έτσι θα αποδείξουμε ότι ε, αν δώσουμε περισσότερη ισχύ και, και ε, όγκο στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και τις κρατικές δαπάνες μειώνουμε και τις ευρωπαϊκές δαπάνες δεν αυξάνουμε. Αυτά ήθελα λίγο να μοιραστώ τα όνειρά μου μαζί σας. Κυρία μου και κύριοι, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε στις παρατηρήσεις που ακούσατε από εκείνους που πήραμε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, βουλευτές που έθεσαν ερωτήσεις ενδιαφέρουσες στις οποίες θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Όπως το είπαν κάποιοι από τους ομιλητές, βασικός στόχος δεν είναι να δημιουργήσουμε περαιτέρω διαιρέσεις. Η προσπάθεια την οποία κάνουμε τα τελευταία χρόνια έχει σαν στόχο την σύγκληση και στον τομέα της άμυνας. Και νομίζω ότι έχουμε καλύψει μια αρκετά μεγάλη διαδρομή τα τελευταία χρόνια. Δεν το κάναμε αυτό εκτός συνθήκης. Πρέπει να κάνουμε όμως τη διάκριση αυτά τα οποία έχουν γίνει μέσα στη συνθήκη και χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και άλλα που γίνονται στα πλαίσια της συνθήκης αλλά δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό. Δεν συμβαδίζουν παράλληλα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη. Είναι λιγάκι δύσκολο έως πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να εξηγήσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη τι ακριβώς συμβαίνει. Καταλαβαίνω λοιπόν τη νομική σας, αν αυστηρότητα, αλλά θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη νομική αντίληψη που ε, δεν εξηγεί το τι κάνουμε. Πρέπει να μιλήσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη με ξεκάθαρη γλώσσα. Φυσικά και θα συμφωνήσω μαζί σας πρόεδρε και σίγουρα η προσπάθεια την οποία κάνουν οι πολιτικοί αυτοί είναι και εμείς εδώ είμαστε για να σας βοηθήσουμε να το πετύχετε. Έχετε λοιπόν το σύνολο της συνεργασίας μου στο βαθμό που σας είναι χρήσιμη βέβαια. Αναφερόμουν σαν παράδειγμα σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει σε επίπεδο διαφρομένης ε, μόνιμη συνεργασία. Άρθρα 46, πρωτόκολλο 10, αλλά οι περισσότερες από τις δράσεις οι οποίες γίνονται στα πλαίσια αυτής της σταθερής ε, συνεργασίας χρηματοδοτούνται και χάρη στις προσπάθειες που έκαναν ε, η Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας όταν δημιουργηθεί με τα ενδιάμεσα μέσα τα οποία έχουν προβλεφθεί αλλά αυτό δεν θα είναι παρά μόνο ένα ποσοστό τελικά. Συστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εργαζόμαστε εκτός συνθήκης ή ε, εργαζόμαστε στο σκότος. Όχι, έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο έχει διευκρινιστεί και υπάρχουν κομμάτια της άμυνας τα οποία χρηματοδοτούνται εκτός προϋπολογισμού. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα άρθρο της συνθήκης το οποίο επιβάλλει όρια το 41 2 το οποίο εμποδίζει την χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό δαπανών που έχουν αποκλειστικά στρατηγική ή αμυντική ε, χρήση. Αυτό είναι ένα άρθρο της συνθήκης το οποίο περιορίζει το τι χρηματοδοτείται από πλευρά του προϋπολογισμού. Ακόμα και στα πλαίσια του άρθρου αυτού βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια ερμηνεία θα έλεγα εφάνταστη και θετική και νομίζω προσπάθησαν να εξαντλήσουν ό,τι μπορούσε να προτείνει η νομική υπηρεσία και πρέπει να το χαιρετήσουμε αυτό γιατί κάτι τέτοιο δεν ίσχυε στο παρελθόν. Έχει υπάρξει πρόοδος. Η πρόοδος μπορεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιητική για όλους αλλά αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα του τελευταία χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εμείνουμε στο θέμα του τρόπου της χρηματοδότησης το θέμα είναι να δούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης για τη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων θα ανήκει στα κράτη-μέλη και θα είναι ευθύνη των κρατών μελών. Αναφερθήκατε στα όνειρα και εγώ μερικές φορές ε, τολμώ να ονειρεύομαι και ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο στο μέλλον θα αυξήσουμε το κομμάτι το οποίο θα χρηματοδοτεί ο κοινοτικό προϋπολογισμός και θα μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε, ας πούμε, να αμφισβητήσουμε ή να αναδιατυπώσουμε το 42. Αλλά τώρα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Και εγώ σαν υπάλληλο στην δική σας υπηρεσία σέβομαι το νομικό πλαίσιο και ε, τα όρια τα οποία δίδουν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ερμηνεία του. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Να πω ότι εμείς εργαζόμαστε στα πλαίσια της συνθήκης όπως έχει τώρα, ως έχει τώρα και οι δράσεις τις οποίες αναλαμβάνουμε ε, εξελίσσονται σε ένα σαφές διαμορφωμένο πλαίσιο προσπαθώντας να πιέσουμε τα όρια όσο μπορούμε πέρα από τις ερμηνείες που κάναμε στο παρελθόν. Ε, υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις και σε σχέση με το 2% του ΑΕΠ. Σαν παράδειγμα το έθεσε και κάποιος από σας η Ευρωπαϊκή Ένωση μήπως ε, συνεισφέρει σε έναν στόχο που δεν είναι στόχος της Ένωσης. Η απάντηση είναι όχι. Η υποχρέωση αυτή είναι μια υποχρέωση των κρατών μελών που ανήκουν στο ΝΑΤΟ και όχι στα υπόλοιπα κράτη. Συνεπώς ε, υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αναλυθεί από όλα τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της ΠΕΣΚΟ, της μόνιμης διαφθομένης συνεργασίας. Έχουν αναλυφθεί λοιπόν κάποιες υποχρεώσεις για την αύξηση των δαπανών και δεν είναι πλέον υποχρέωση του ΝΑΤΟ μόνο, αλλά υποχρέωση και των κρατών μελών της Ένωσης. Και αυτό το οποίο κάνουμε στην παρούσα φάση είναι να εργαζόμαστε πάντα στο νέο αυτό πλαίσιο. Υπήρξαν επίσης και αρκετές ερωτήσεις για την κινητικότητα. Η κινητικότητα και την διπλή χρήση, η διτή χρήση. Εμείς στα πλαίσια της κινητικότητας χρησιμοποιούμε την δυνατότητα που μα δίνει η διτή χρήση. Η διαδικασία για την κινητικότητα στην παρούσα φάση είναι καταρχάς η προσπάθεια ανείχνευσης, εντοπισμού ε, των στρατηγικών στρατιωτικών μεταφορών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες του, αλλά είναι μια προσπάθεια την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία προσπαθεί να καθορίσει τις ανάγκες σε επίπεδο υποδομών οι οποίες θα πρέπει να συμφωνηθούν σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσει μια διαδικασία εντοπισμού των προγραμμάτων τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα μέσα τα οποία θα θέσει στη διάθεσή μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά γίνονται επί τη βάση των λεγόμενων μέσων διπλής χρήσης. Δεν θα γίνουν προσπάθειες μόνο ε, για να βοηθηθούν οι στρατιωτικές μεταφορές, αλλά και οι μεταφορές ε, ε, κανονικής χρήσης, μη στρατιωτικής χρήσης. Η διαδικασία λοιπόν στην οποία μπαίνουμε τώρα για την κινητικότητα, την στρατιωτική, είναι κάτι το οποίο εσείς γνωρίζετε, είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τις ανάγκες φυσικά υποδομών, υπάρχουν θέματα κανονισμών, υπάρχουν θέματα νομικά, υπάρχουν θέματα τελωνιακά, υπάρχουν θέματα αδειοδοτήσεων, Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια των προσπαθειών οι οποίες θα γίνουν τους επόμενους μήνες για τη διευκόλυνση των μεταφορών αυτών. Υπάρχουν λοιπόν θέματα που άπτονται των υποδομών, υπάρχουν όμως και θέματα που άπτονται ε, της νομικής φύσης των ρυθμίσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τους σχετικούς κανονισμούς. Πρόκειται λοιπόν για μια τεράστια προσπάθεια την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ωφελήσει όμως και το ΝΑΤΟ το οποίο ο ΝΑΤΟ από μόνο του δεν είναι σε θέση να το κάνει. Εμείς λοιπόν το κάνουμε και για το ΝΑΤΟ αλλά και για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Συνεπώς λοιπόν δεν ξέρω αν έχετε και άλλες ερωτήσεις αλλά νομίζω ότι απάντησα. Δυστυχώς ε, η συζήτηση ναι μεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ε. Ο κύριος Πρέζα, κάποιες ευθυνήσεις και συμπληρώσεις. Κυρία Τωμά, ναι, όντως, τρία κράτη πρέπει να συμμετέχουν. Ζητώ συγγνώμη αν είπα δύο ε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου. Εγώ έκανα Ε, θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω το εξής. Τα 6,5 δισεκατομμύρια για τις αρτιωτικές μεταφορές έρχονται να προσθεθούν ε, στη ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτά είναι χρήματα που προστίθενται, δεν είναι ότι έχουμε περικοπές, εκτός από την ε, χρήση. Ε, τώρα για την ενότητα του προπολογισμού και τη διάρθρωση του προπολογισμού ε, θα συμφωνήσουμε εύκολα, δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτό. Και στις προτάσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης να εγγραφεί στον προπολογισμό. Ναι, βεβαίως. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα τμήμα που αντιστοιχεί και σε στρατιωτικές δράσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και θα κληθούμε να το διαχειριστούμε. Και όπως είπε και, ε, ε, και ο κύριος Σεράνος προηγουμένως, εμείς ε, εργαζόμαστε χωρίς τροποποίηση των συνθήκων με τις συνθήκες όσες έχουν αυτή τη στιγμή. Μιλήσατε για τις ε, προμήθειες οπλικών συστημάτων και τι αγοράζουν τα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνουμε ένα σύστημα για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και τα αντίστοιχα κονδύλια. Ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να ενθαρρύνουμε και τα κοινά προγράμματα, αλλά να ενθαρρύνουμε και να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε και μια στρατηγική αυτονομία ακριβώς και αφορά και τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Ευχαριστώ. Κυρία Χάρδεμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι με κάλυψαν και δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το συμπέρασμα θα μας το δώσει η κυρία Μούντι. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές για τις λεπτομερείς παρουσιάσεις και τις απαντήσεις που δώσατε στα ερωτήματα. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για πολύ ακόμα, να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα της κυβέρνηση την ε, ενότητα προς τον προϋπολογισμό. Όμως, θεωρώ ότι η δέσμευση και των δύο επιτροπών αναδεικνύει τη σημασία του θέματος και το πόσο ε, σοβαρή απόψη το λαμβάνουμε το θέμα. Θα είναι ένας συνεχιζόμενος αυτός ο διάλογος μεταξύ μας και μεταξύ σας και βλέπουμε και το χρονοδιάγραμμα πώς θα προχωρήσουμε στην νομοθετική διαδικασία και τα βήματα που θα λάβουμε για το επόμενο πολιετές δημοσιομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την κοινή συνεδρίαση όπου μας δόθηκε ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Merci, Claire. Ευχαριστώ, Claire. Σας ευχαριστώ κυρία μου και κύριοι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ Κλέα.